καλή εκπροσώπηση, γιατί αυτή η συνεδρίαση ήταν ε, απαραίτητη. Έχουμε κάποιες ειδικές αποφάσεις στο Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε. Θα ήθελα να εγκρίνουμε την ημερήσια διατάξη, η οποία είναι πάρα πολύ σύντομη σήμερα. Ελπίζω να μην έχετε οποιαδήποτε επιθυμία να αλλάξει η ημερήσια διατάξη. Όχι, ωραία, άρα εγκρίνεται λοιπόν η ημερήσια διατάξη. Έχουμε τις ανακοινώσεις της Προέδρου. Σήμερα διατίθενται όλες, ε, όλες οι γλώσσες για διερμηνία, εκτός από εσθονικά και μαλτέζικα, για τους τριμερείς διαλόγους τώρα. Να σας κάνω μία σύντομη παρουσίαση του πώς έχουν τα πράγματα στον τριμερή διάλογο. Ο τριμερής διάλογος ε, ασχολείται με τις ε, πρόσβαση και στις γενετικούς πόρους και τη σωστή χρήση και διανομή, αν θέλετε, των ωφέλων σε ό,τι αφορά και την ε, βιολογική ποικιλότητα. Τρεις ε, τρίλογοι έλαβαν χώρα. Στις 28 Νοεμβρίου θα λάβει χώρα ο τρίτος τριμερής διάλογος στις 6.30 ύστερα. Έχουμε την έκθεση Ότσκι για το επίπεδο εκπομπής θορύβου των ε, οχημάτων. 5 Νοεμβρίου έγινε μια συνεδρίαση στα πλαίσια τριμερούς διαλόγου. Έχουμε τα κλινικά πειράματα επίση, τριμερού διαλόγου. Χτε το βράδυ έλαβε χώρα ένα ε, τέτοιο τριμερή διάλογο, Γκλένι Βίλμουτ και έχουμε προβλέπονται άλλε δύο συνεδριάσει ε, τριμερούς διαλόγου. Ελπίζουμε μήπω και πετύχουμε συμφωνία στην επόμενη συνάντηση, αλλά είναι δύσκολο το θέμα σίγουρα. Οι τριμερείς διάλογοι προβλέπονται και για την, ε, το πρώτο ήμιση του Δεκεμβρίου. Επίσης έχουμε ε, την έκθεση για τα θωρεούχα αέρια. Αυτές λοιπόν είναι οι ανακοινώσεις. Ελπίζω και αυτοί οι τριμερείς διάλογοι να μπορέσουν να συνεχιστούν σωστά. Για σήμερα έχουμε ένα σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η ψηφοφορία για την έκθεση για την τροποποίηση ορισμένων οδηγιών στον τομέα του περιβάλλοντος, της γεωργία, της κοινωνικής πολιτικής και της δημόσιας υγείας λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ένωσης. Όπως σας ανέφερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η Μαγιώτα θα πρέπει να είναι υπερπόντιο διαμέρισμα και γι' αυτό λοιπόν ε, θα πρέπει να τηρήσουμε τα σχετικά χρονοδιαγράμματα. Γι' αυτό και μας κάλεσαν σήμερα το πρωί να ψηφίσουμε επί της έκθεσης αυτής. Ο κύριος Γκρότε είναι ο εισηγητής, ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο οποίος δυστυχώς ε, δεν μπορεί να παρευρεθεί. Θα ήθελα να παρακαλώ να σας ζητήσω την κατανόησή σας. Είναι η πρώτη ε, ψηφοφορία την οποία προεδρεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για την κατανόησή σα και για τη βοήθειά σας. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Διαπιστώνω λοιπόν ότι είμαστε αρκετοί. Διαδικαστικό, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια και πιεζόμαστε, ε, ε, έχουμε, έχουμε επαρκή αριθμό παρών των βουλευτών. Απαρτία υπάρχει. Ναι, κοιτάξτε, θα πρέπει να είμαστε 18 και είμαστε περίπου 20. Είμαστε αρκετοί λοιπόν. Λοιπόν, να ψηφίσουμε. Να ξεκινήσουμε με την τροπολογία 9. Και ρεγγιένα. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Περνάμε Στο άρθρο 1, τροπολογία 2 και 13. Υπέρ. Κατά. Άρθρο 1, άρθρο 1 λέει ο Πρόεδρος. Τροπολογία 2 για το άρθρο 1 και 13 για το άρθρο 1. Also, Ψηφίζουμε από κοινού την τροπολογία 2 και την 13 και την 4 της Επιτροπής Ρέγγι. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Καταπίπτει. Και ψηφίζουμε την 5 της Ρέγγι. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 καταπίπτει. Η 6 της Ρέγγι. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. οι 15 και οι 5. Ταυτόσιμες. Και οι 7 της Ρέγγι. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Στη δεύτερη παύλα. Υπέρ, κατά, Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε παρακαλώ, να κάνουμε έναν ηλεκτρολικό έλεγχο για την τροπολογία υπερθυμών 15. Πέρας ψηφοφορίας. 24 ψήφοι. Συνολικά 12 υπέρ, 12 κατά, άρα απορρίπτεται. Και περνάμε λοιπόν στην 6 και ρέγγι 8. Υπέρ. Κατά. εγκρίνεται Τροπολογία 7 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα, η 16 στο δεύτερο τμήμα της παρακαλώ υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 8. Καταπίπτει. Και σε ό,τι αφορά την 9 επίσης ε, καταπίπτει. Οι άλλες τροπολογίες λοιπόν έχουν ήδη ψηφιστεί. Και περνάμε στην τροπολογία 21. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνουμε μια τεχνική προφορική τροπολογία. Σας είπα προηγουμένως ότι ε, από την 1η Ιανουαρίου θα τεθεί σε ισχύ και θα τα ψηφίσουμε αυτά στην Ολομέλη του Δεκεμβρίου. Ενδεχομένως να υπάρξει πρόβλημα λοιπόν αν υπάρχουν μόνο 20 μέρες για να τεθεί σε εφαρμογή. Γι' αυτό θέλω να κάνω την προφορική τροπολογία να διαγραφεί το σε 20 ημέρες. Η οδηγία λοιπόν, θα λέει το κείμενο, θα τεθεί σε ισχύ από την δημοσίευση της στην επίσημη εφημερίδα της κυβερνήσεων και θα ισχύει από 1η Ιανουαρίου. Αν είσαστε λοιπόν υπέρ της προφορικής τροπολογίας αυτής, παρακαλώ ψηφίστε υπέρ. Υπέρ λέω. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Στις τελογικές σκέψεις, 10, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οι δύο της Ρέγγι. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τρία της Ρέγγι υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 καταπίπτει και περνάμε λοιπόν στην τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιος είναι υπέρ της τροποποιημένης πρότασης έναξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Αν ψήφισατε όλοι, ολοκληρώθηκε έτσι η ψηφοφορία. 24 ψήφοι, 17 υπέρ, 6 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν η, το τοποποιημένο κείμενο και τώρα θα ψηφίσουμε το νομοθετικό ψήφισμα. Έναρξη ψηφοφορία, παρακαλώ. Αν ψηφίσατε όλοι, πέρα ψηφοφορία. 23 ψήφοι λέει ο 20 υπέρ, καμία κατά, καμία αποχή. Συνάδελφοι, εγκρίνεται λοιπόν η έκθεση και έτσι μπορεί να συνεχιστεί η ροή των εργασιών. Σας ευχαριστώ ειλικρινά. Σας ευχαριστώ και για την υποστήριξή σας, για την ταχύτητα της ψηφοφορίας και ολοκληρώνεται έτσι η συνεδρίαση. 27 Νοεμβρίου η επόμενη συνεδρίαση στις 9 το πρωί μέχρι τις 12.30. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τη γραμματεία σας. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας.